Good uh, morning, uh, everybody. Ε, καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ορίσατε στην τελευταία συνεδρίαση. Break, uh, στην τελευταία συνεδρίαση πριν τις εννέες διακοπές, όπως βλέπετε είναι αμυγός ψηφοφορία. Ε, τρία θέματα έχουμε να ψηφίσουμε. Ε, μου ζητήθηκε να αλλάξω λίγο τη σειρά των ψηφοφοριών. Άρα θα ψηφίσουμε πρώτα την εντολή που αφορά ε, την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που έχουν την ευθύνη για την επιβολή της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Um, where, um, the is... Η συγκήτρια είναι η κυρία Σενάλοβα Παρακαλώ, δεν ξέρω αν θέλετε το λόγο. Δεν θέλετε. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να ε, περάσουμε αμέσως στη ψηφοφορία που είναι μία και μοναδική ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα. Πέρας, εάν ψηφίσατε όλοι φυσικά, όχι δεν έχει κλείσει ακόμα. Από ό,τι φαίνεται, ε, ένας δεν έχει ψηφίσει ακόμα, πέρας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια, κυρία Σένα Λοβά. Okay. Ωραία. Ε, σημαίνει τώρα αυτό ότι ε, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο κατάλογος. Είναι το θέμα η διάθεση προϊόντων λίπανσης και η συγγήτρια είναι η κυρία Γκάλ Πέλτς. Θέλετε το λόγο. Α, μετά την ψηφοφορία. Ωραία. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Μπορούμε να περάσουμε τώρα μέσω στην ψηφοφορία. Και θα ψηφίσουμε πρώτα Τη συμβιβαστική 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 86 87 και η ένα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τι είναι αυτές, ταυτίζονται μεταξύ τους. Μάλιστα, είναι ταυτόσημες. Ε, ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. απορρίπτω τέτε το σύνολο ένα της Επιτροπής Γεωργίας ως προσθήκη ψηφί παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία υπαριθμών 18 ψηφί κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ όχι, 156 πρώτα. Ωραία. Μάλιστα. 156 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. Η 157, 158 και NV15 μαζί. Είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω αυτό θέλει έλεγχο. Μπορούμε να την ελέγξουμε αυτή την ψηφοφορία σας παρακαλώ. Αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, άγκρι 23, 159, 160 και NV 16. Ψηφίπε κατά αποχές εγκρίνεται. Το είναι η τροπολογία 161 162 άγκρι 24 και ένβι 17 όλες μαζί ψηφίπε κατά άποχες αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ close Πέρασε. Απορρίπτεται. Ωραία. Ε, συμβαστική 16. Ψηφιπέ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 169 μαζί με την 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στη συνέχεια Αλλάζουμε σελίδα. Οι τροπολογίες 172, 173, ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω και εδώ χρειάζεται επαλήθευση. Παρακαλώ. Vote closed. And it's adopted. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 174 Είπε. κατά, αποχές απορρίπτεται η τροπολογία παρθμών 20 ψήφιπε, κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 21 υπέρ κατά απόχες Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Μπορούμε να την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 21, πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν εβδομήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω θα πρέπει να την ελέγξουμε και αυτή. Vote is closed. Εγκρίνεται. 22, 178, 179 και 180 υπέρ. Είναι ταυτόχρονα κατά. Απόχες. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. 181, άγκρι 30, NV 20, ταυτόσυνες ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία 183, ψηφιπέρ κατά αποχές. Εδώ νομίζω χρειάζεται έλεγχος, αρχίζει η ηλεκτρονική απολύτευση. The vote is closed. Ah, it's rejected. Α, περίφθη. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε την 184 ψηφιπέ κατά αποφυγές απορρίπτεται 182 μαζί με τη 212 239 ε, και 135 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. 185 μαζί με την 195 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 17 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 24, 189, 190, 191 και 192. Όλες αυτές ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 18 υπέρ. Against abstentions. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 20 υπέρ. Α, μαζί με τη συμβαστική 24 και τη συμβαστική 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Η ε, τροπολογία 201 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 202 μαζί με 230 και 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 24 υπέρ, 25 συγγνώμη, κατά αποχές. Νομίζω χρειάζεται παλήθευση και αυτό. Αρχίζει ψηφοφορία για την τροπολογία 25. Πέρας. Εγκρίνεται. 204 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 31 υπέρ. Κατά. Α, okay. Α, μάλιστα. Εγκρίθηκε 204, οπότε καταπίπτει 31 της Επιτροπής Γεωργίας και προχωρούμε στην τροπολογία 27 ως προσθήκη. Ψηφί υπέρ. Κατά. 27. Είμαστε στην 27. Ο κύριος Ταραμπελά ζητεί το λόγο. Yeah, we have to vote, apparently. Μα πρέπει να την ψηφίσουμε. Μάρκ, ε, θα ήθελα να πω το εξής. Ψηφίσαμε την τροπολογία 31 της Επιτροπής Γεωργίας, η οποία καταπίπτει σε περίπτωση που εγκριθούν οι 203 και οι 204. Όχι η μία ή η άλλη, αλλά η 203 απερίφθη της κυρίας Μέιμπελ. So ah. ah, we don't have to Yes. Donc, Μήπως να βάλουμε αν εγκριθεί 203 ή 204. Είτε η μία είτε η άλλη, όχι και οι δύο. Αλλιώ καταπέπτει. Μάλιστα, για να το καταλάβουμε. Ωραία. Είμαστε στην τροπολογία 27. Δεν την ψηφίσαμε αυτή falls. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to amendments. 27 λοιπόν. Ο κύριος Κοέγιο. 27 ε, Λέει, λέει ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί γιατί σχετίζεται με την 23. Μάλιστα, ωραία. Ε, πάμε στη 210. Υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει πορευθεί. Όχι, ας το ελέγξουμε παρακαλώ. close vote. adopted. Μάλιστα εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβιβαστική 22, ψηφί Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Α, όχι, δεν ψηφίζουμε. Την έχουμε ψηφίσει. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. η τροπολογία 30, το πρώτο τμήμα, ψηφίπε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία συμβιβαστική, 26, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί, τη ψηφίσαμε και προχωρούμε στην τροπολογία 34, βλέπω εδώ. Ψηφίπε, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 35 τώρα είπε. Όχι, έχει 2,47 πριν. 247. Okay. Ε, Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι θέλει έλεγχο αυτό. Την 247 παρακαλώ. Thank you. We close the Πέρας. Εγκρίνεται. Α, τώρα θα ψηφίσουμε την 35. Όχι, διότι καταπέπτει. Επειδή εγκρίθηκε η 2.47. Γι' αυτό έπρεπε να ψηφίσουμε πρώτα τη 2.47 και μετά τη 35. Συμβαστική 27. Ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 251. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 37 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Μπορούμε να την ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρας; Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 μαζί με τις συμβαστικές 44 και 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία 260 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 39 μαζί με τις 40, 41 και 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 241 σύμβατη με την 39 ψηφίπε κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε. Η τροπολογία 263 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 271 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 272 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 273 μαζί με την 44 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 31 υπέρ είναι μαζί με τη συμβαστική 5, 14 και την M38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Προχωρούμε στην τροπολογία 291. Ψηφί υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται. Τσεκ φωνές. Ας την ελέγξουμε. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί. We close the vote. Πέρας. Αχ, Μάρκ. Αν είχαμε βάλει στοίχημα θα είχες χάσει. Απερίφθη. Συμβαστική 32 μαζί με την 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική την 33 μόλις την ψηφίσαμε. So we go to amendment 3. Η 302 ψηφίπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 303 και NV34 ε, ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται we adopted 304, so this 305 falls. Okay. So we go down to um, Okay, we can move to Agri 30. Agri 39 μάλλον πρέπει να πάμε γιατί τα άλλα έχουν καλυφθεί. Ε, υπέρ της τροπολογίας 39 της Επιτροπής Γεωργίας κατά αποχές. Νομίζω ότι χρειάζεται επαλήθευση και αυτό παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία για την Άγκρη 39. Απορρίπτεται. Συμβαστική 34 μπλοκ με την 49, 50, 51, 15, 474 και άγρια 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια συμβαστική 36 μπλοκ με την 51 και την ίντα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 συμβατή με την 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται εντάξει δεν είπα τίποτα μετά έχουμε την τροπολογία 321 ως προσθήκη είπε κατά αποχές απορρίπτεται 322 έχει αποσυρθεί 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 324 και άγκρι 41 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 325 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 326-327 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. NV 40 καταπίπτει. Άγκρι 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκε 3.25, οπότε η άγκρη 43 καταπίπτει και πάμε στην 3.28. Είπε... 3.29 συγγνώμη, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Then we move to Agri 45. Uh, uh, uh, Agri. we have to vote on 333? Okay. So we have to... Λοιπόν, την 333 πρέπει να ψηφίσουμε ως προσθήκη πάντα. Τη βρήκατε λίγο πιο κάτω. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα η Άγκρη 45 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Μπορούμε παρακαλώ να την ελέγξουμε. Άγκρι 45. The vote is closed. Πέρα συγκρίνεται. 3.34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. Συμβιβαστική 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. «54» είναι με την έμβη 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένβι 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 344, 345 και άγκρι 49. Πάμε στην 52, άγκρι 52, υπέρ, κατά, εγκρίνεται 351 352 υπέρ κατά αποχές είναι ταυτόσιμες παρόλα αυτά να το δούμε ηλεκτρονικά 351 και 352 μαζί ηλεκτρονικά παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας Ώρα, λοιπόν εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άγκρι 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές. Λοιπόν, στην έμβη 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 353 και άγκρι 52 μαζί, α, καταπίπτουν. 355 υπέρ, κατά, αποχές. Και εδώ θέλω να το δούμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, την 355 παρακαλώ να ψηφίσουμε. Εγκρίνεται. 357 και άγκρι 53 με υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω εγκρίνεται. 358 που είναι συμβατή με την 357 και την άγκρη 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 359 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 360-361 είναι ταυτοσμης υπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην άγκρη 56 άγκρη 56 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 366 367 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV Άγκρι 58 υπέρ κατά αποχές ε, εδώ νομίζω πρέπει να το δούμε ηλεκτρονικά Άγκρι 58 παρακαλώ πολύ πέρας εγκρίνεται 368 και άγκρι 59 ταυτόσπιση υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 369, 369 με συγχωρείτε, υπέρ. Α, θέλετε να δούμε το άγκρι 60, ωραία, την τροπολογία αυτή ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά, άγκρι 60. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 369 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 370 και άγκρι 61 μαζί ταυτόσμες υπέρ, κατά, αποχές. Και εδώ θέλω ηλεκτρονικά παρακαλώ να ελέγξουμε την 370 και άγκρι 61. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 55 υπέρ, κατά, αποχές

θα πρέπει να ψηφίσουμε και την 379, τροπολογία 379. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 379. Το βρήκατε? Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Μπορούμε να το κοιτάξουμε και ηλεκτρονικά στην 379, πρώτο τμήμα. Παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 43, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 57. Με την 411 και 412 με ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην 454 που είναι ε, ταυτόσιμη με την έμβη 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV73 και Άγκρι 91 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Άγκρι 92 υπέρ. Κατά. Αποχές και νομίζω απορρίπτεται. Θέλω να δούμε ηλεκτρονικά την Άγκρι 92. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 456-457 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά nv 79 είναι ε, σε βλοκ είναι με την nv 115, οπότε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν η 459, οπότε περνάμε στη συμβιβαστική 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 44 και εδώ unblock για την άγκρη 99 διαβάστε τα υπέρ κατά αποχές νομίζω εδώ πρέπει να το δούμε άγκρη 99 ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται Μετά 462 υπέρ. Κατά. Άποχες. Παρακαλώ. Να σηκώσετε τα χέρια σας για την 462 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτετε 463 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 465 υπέρ κατά αποχές εδώ δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για την 465 σας παρακαλώ πολύ ηλεκτρονικά Close the vote. It's rejected. Απορρίπτεται λοιπόν. Άγκρι 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 466 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 112 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 113 άγκρι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. NV 98 υπέρ, συγγνώμη 89, NV 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να το δούμε. Για να, εξετα... Για να δούμε λοιπόν ηλεκτρονικά την MV89. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άγκρι 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 469 που είναι η Άγκρη 116 και 98 έμβη που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 470 και έμβη 99 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 118 υπέρ, α, ε, ε με την 119 και 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θα το δούμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Λοιπόν, άκρη 118. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ίντα 4 υπέρ, κατά, αποχές και νομίζω εγκρίνεται. Θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την ίντα 4. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 4,71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβι... Όχι. 4,72 υπέρ. Κατά. Απο... Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4,73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 482 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 άγκρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 483 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 484 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην άγκρη 135 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 136 άγκρη υπέρ. Άγκρη 136 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Νομίζω να κάνουμε μία ηλεκτρονική επαλήθευση την άγκρη 136. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε μετά στην 485 και 137 άγκρι ταυτόσιμες, αμπλοκ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην 486 με την m 103 Γιατί, λέει η πρόεδρος. Ωραία λοιπόν. Περνάμε στην άγκρη 138. Άγκρη 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 έμβη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά περνάμε Ένβη 106. Συγγνώμη, στην 105. Ένβη 105 εμπλοκ ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμβη 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άγρι 143 υπέρ εμπλοκ πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άγρι 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε να το δούμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, είναι προφανές. Η άγρια 149 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένβια 109, αμπλόκ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 άγκρι υπέρ, κατά, κατά, αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 156 unblock υπέρ άγκρι. Τι κάνουν οι σοσιαλιστές. Υπέρ, κατά, αποχές. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ηλεκτρονικά την άγκρι 156. We close the vote. It's rejected, so it's one uh, vote. Then, uh... Απορρίπτεται. 489 <laughs> και 490 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 491 και 1,112 112 καταπίπτουν. Α, καταπίπτουν. 492 ε, και 493 και 494. Ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 495 άγκρι 159 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά, αποχές, Νομίζω δεν εγκρίνονται, αλλά να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. 4,96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 1.13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει. 196. 4.96. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 165 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται. Ένβη 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές έλεγχο. Ελέγχουμε την 45. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 5.51 και 5.52 πανομοιότυπες. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Άγκρι 167 513 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβη 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 167 Ένβη 122 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άγκρι 167, έμβη 122. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Άγκρι 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 και 514 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 516 και 169 της Άγκρη κατά αποχές εγκρίνεται 557 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 518 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 519 και 520 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 551-552 521-522 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 525 άγκρι 171 ταυτόσημες unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 526 και άγκρι 172 Α, ωραία, καταπίπτει 523, 524, 527 7 unblock υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Άγκρη 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 529 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Να ελέγξουμε 529 Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 123 της ΕΝΒΗ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 533, 532, α, καταπίπτουν. 503 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 535 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρι... απορρίπτεται. 124 της ΕΝΒΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 της ΕΝΒΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 539-540 καταπίπτουν. 544, 545, 546 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 547 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 548 και άγκρι 178 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 549 και 470 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 550 και 180 της άγκρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ελέγξουμε πέρας Εγκρίνεται. Άγκρι 182 και 551 και 552 ταυτόσημες. 551 μόνο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 552 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 553 κατά πίπτη... 555 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν 557 έγκρι 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 558 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική 52 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 566 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 566 567 και 568 ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 569 μπλοκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω 569 να ελέγξουμε απορρίπτεται 570 και 571, άγκρι 192 ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ένβι 180 υπέρ 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ 573, 574, 575 και 576 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε, 577, 78, 79 πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 586 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 588 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «588 υπέρ κατά αποχές, ε, ε, κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο μάλλον. Δίκιο είχατε που ζητούσατε έλεγχο. Άγκρι 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 της Άγκρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μάρκ. Με συγχωρείτε πρόεδρε να πάω πίσω. Σελίδα 56. 126 της Ένβη. Δεν ψηφίστηκε. Ενώ η δική μου 529 απορρίφθηκε. Οπότε δεν κατέπιπτε η 126 της Ένβη. Εκτός και αν έχω καταλάβει λάθος. 529 απορρίφθηκε, από ό,τι κατάλαβα. Θα έπρεπε λοιπόν να ψηφίσουμε την ένδια 126, αλλά δεν ψηφίστηκε. ...126 μάρκα. But it is, so it, it followed. No, is it five six, five? So we have to that one. one yes, we have to. One six. And we want to six, yes. six. we have to, yes. I think, I think you're right, Mark. In Page Non, c'est Madame Pocky, Sarah c'est notre η κυρία Σάρα Πόκη που είναι συμβουλός μας εδώ μου το υποσημείωσε. Εγώ ήμουν στη Παρεσυρμένο από τη δράση. Ναι, NV 126 πρέπει να την ψηφίσουμε. Την έχετε βρει εντωμεταξύ. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Sorry, Mark. Απορρίφθηκε. Να τσεκάρουμε και κάτι άλλο. We need to check um, apparently amendment 174. 174. 174. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 174. 74. Ποιος θα τη βρει πρώτη, πρώτος σε, αυτή την, ε, σε αυτόν τον κατάλογο. Page 55 in the socialist list. No, it's not 174, it's 74. Όχι 174, 74. 74. I found it. Εγώ το βρήκα. Σελίδα 54. Ταυτόσιμη με την 514. Το βρήκατε όλοι υπέρ, κατά. Περιμένω τους σοσιαλιστές. Ψηφίζουμε την 7-4.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 actually 30, and then the 20 were adopted. That so is the correction. So so it's fair. yeah. Okay, so um, normally uh, we adopted 70. Λοιπόν, οι 74 και 145 εγκρίθηκαν, αλλά είχαν καταπέσει, διότι εγκρίναμε τις τροπολογίες 181 και την NV20. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε τίποτα, από όσο έπρεπε να το ανακοινώσω όλο αυτό. Okay. Okay. And now we move to... Can we check the... Να ελέγξουμε την άγκρη 166. 166 μπορούμε να την ελέγξουμε. Madame, excusez-moi, mais il y a une confusion. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ της NV74 σελίδα 40 στον κατάλογό μου ή της 74 που δεν είναι εύδυνδη της σελίδας 53. Ε, Αυτήν πως δεν ψηφίσαμε. Κανένα από τα δύο. Όχι, ήταν απλώς μια αναγγελία πρέπει να την κάνω. Η κυρία Γκάλ Πέλτ ζητά να ε, ελέγξουμε για την τροπολογία Άγκρι 166. 166. Okay, it was adopted. Εγκρίθηκε γιατί 551 και 552 απορρίφθηκαν. Όχι, τώρα εντάξει είμαστε. Προχωράμε. Συμβιβαστική 2. Είμαστε σχεδόν στο τέλος. Συμβιβαστική 2 στις ιδεολογικές σκέψεις. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, όχι, εγκρίνεται. Με συγχωρείτε, Μάρκ. Συγγνώμη. Πω, πω, συγγνώμη. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία να ελέγξουμε. Πέρας, εγκρίνεται. NV4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 ταυτόσιμη με την 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 15, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104, 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151-152 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται απορρίπτονται 13 της ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. I close Πέρας αυτής και εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στον εισηγητή την εισηγητρία. Ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την τεράστια αυτή ε, δουλειά που κάναμε. Πρώτα τους και την κυρία Γκαρντίνη, τον Μάρισλαβ και όλους τους συνεργάτες φυσικά που επιτέλεσαν ένα ε, ε, ηρωικό κυριολεκτικά έργο. Και φυσικά τη γραμματεία όλους ιδιαιτέρως. Αυτή είναι η έκθεση. Θα μπορούσα να συνεχίσω τις ευχαριστίες. Είναι μακρύς ο κατάλογος των ανθρώπων που δούλεψαν, που αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο και κόπο. Στην αρχή απήχαν πάρα πολύ οι θέσεις μας. Ε, στη συνέχεια πλησίασαν μεταξύ τους. Υπήρξαν πάρα πολλές τροπολογίες και επιτέλους εγκρίναμε την έκθεση. Ελπίζω τώρα η Εστονική Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί για να εγκριθεί και στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αυτής. Η νομοθεσία αυτή ε, θα μειώσει ε, και το γραφειοκρατικό ε, άχθος για τις επιχειρήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. με τη μείωση αυτή της γραφειοκρατίας και ε, τις ενιαίες ρυθμίσεις που προβλέπονται διευκολύνεται πολύ η ζωή τους. Τώρα όμως υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Υπάρχει μια ρήτρα που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί ε, όλη αυτή την εφαρμογή στην πράξη ως προς την εναρμόνιση και την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ελπίζω το συγκεκριμένο πακέτο να αποτελέσει ένα λιθαράκι για την κυκλική οικονομία και για την ε, κυκλοφορία στην αγορά νέων καινοτόμων προϊόντων. Είναι η τελευταία συνεδρίαση στην οποία συμμετέχω. Σας εύχομαι ό,τι υποθείτε για το μέλλον και καλή δουλειά στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για όλη αυτή τη σκληρή δουλειά και φυσικά εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ, 3 ακάτα και μία εποχή. Μάρκ Ταραμπελά θέλει να πάρει το λόγο. Ε, Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής. Υποθέτω ότι όλοι οι σκιώδεις θα συμφωνήσουν μαζί μου για να ευχαριστήσουμε την κυρία Γκάλ Πέλτ για το επικοδομητικό της ε, πνεύμα. Ήταν δύσκολο το θέμα τεχνικό με αποκλίνουσες απόψεις. Προσπάθησε να βρει συμβαστικές προτάσεις και δεν ήταν καθόλου εύκολη η δουλειά αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη γραμματεία και εσείς κυρία Συγήτρια το κάνατε, τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων, ε, τους υπαλλήλου μας, τους βοηθούς μας. Είναι η τελευταία φορά ε, ε, που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει καθήκοντα από άλλο μετερίζει. Εμείς την ψηφίσαμε να πάει εκεί. Ε, πάντως θα χάσουμε ένα αξιόλογο στέλεχος με επικοδομητικό πνεύμα. Θα πρέπει να τη χειροκροτήσουμε, το αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ και να ε, είναι ούριος ο άνεμος στη νέα σας θέση. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι. Καλή τύχη στα επόμενα καθήκοντά σας και στην υπόλοιπη σταδιοδρομία σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό μας φέρνει την τελευταία ψηφοφορία τώρα για σήμερα, που είναι ο Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2018. Η συγκητής είναι ο Ντάν Ντάλτον. Θέλεις το λόγο, ο Ντάν. You want to take the floor Θέλεις το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που απέσυραν τις τροπολογίες μετά τις αξιολογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά. Πάμε λοιπόν στη ψηφοφορία. Ας προχωρήσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε πρώτα ε, τη γνωμοδότηση. Ε, η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ, κατά,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 αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε, αρχική ψηφοφορία. I close close the vote. Πέρας. 30 ψηφί υπέρ, 4 κατά χωρίς αποχές. Και τώρα θα ψηφίσουμε ε, τις γραμμές στο προπολογισμού. Ε, Badge 1. Χωρίς σχόλια. Για να επανέλθει το κονδύλι του σχεδίου προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε στην τροπολογία Badge 6. Πρώτα τα σχόλια. Ψηφί κατά αποχές εγκρίνεται. Και στη συνέχεια ε, τα ποσά, ψηφίπε, συγγνώμη, ο κύριος Στέφανετς. Και τα σχόλια του budget 2 πρέπει να ψηφίσουμε. Okay, okay. Thank you ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Όντως, καλά που μου το θυμήσατε. Θα πρέπει να ψηφίσουμε το IMCO Badge 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα τα σχόλια μόνο στη budget 3. Η 3 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Εντάξει, μόνο τα σχόλια είπαμε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα Τα ποσά για το 6, τα σχόλια τα ψηφίσαμε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, Badge 7, τα σχόλια, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τα ποσά τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 8 έχει αποσυρθεί, η 9 τα σχόλια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τα ποσά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μάρκ νομίζω ότι θα σε πυροβολήσω τέτοια εντύπωση σου δίνω Α. τα σχόλια ημκομπάτς 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα ποσά υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ΥΜΚΟΜΠΑΤΣ 11, τα σχόλια υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, τα ποσά υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. ΥΜΚΟΜΠΑΤΣ 12, έχει αποσυρθεί, άρα τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι είμαστε στο τέλος, χαρητήρα κύριε Σιγητά, εγκρίθηκε η ε, πρότασή σας κύριε Ντάλτον. Θέλετε να πείτε τίποτα τώρα. Πάρα πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους μας για την υποστήριξη. Έχουμε μια πολύ καλή βάση προτάσεων και τίποτα από αυτά που προτείνουμε δεν είναι εξωφρενικά. Άρα ε, ελπίζω να ευδοκιμήσει αυτή η πρόταση. Εμείς θα την υπερασπιστούμε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την υπομονή σας. Ήταν περίπλοκη η ψηφοφορία και οι λίστες. Για μένα πρώτη φορά κάνω ψηφοφορίες. Ε, ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίασή μας. Η επόμενη θα ε, διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία σας σε αυτή την κοινοβουλευτική χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και τη γραμματεία τους συναδέλφους μου φυσικά ευρωβουλευτές και πάνω απ' όλα και το σημαντικότερο, καλές διακοπές σε όλους σας. Για να επιστρέψετε με πολύ δυναμισμό. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε. Thank you very much.